Allora, possiamo iniziare. Ο Πρόεδρος, λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε και να σας πω πρώτα-πρώτα τις ανακοινώσεις, αυτά τα οποία αποφασίστηκαν από τους ε, συντονιστές οι οποίοι συνεδρίασαν. Μιλήσουμε. Θα τα πω μετά την ψηφορία για μην φύγετε, οπότε ξεκινήσουμε τώρα όσον αφορά την ε, ε, ψηφοφορία για την ε, σύνδεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιση των εκλογών. Παράγραφος 2, τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ, σηκώ στα χέρια, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επομένως, καταπίπτουν η 16, α, όχι, 16, μόνο η 16 λέει ο πρόεδρος και τώρα πάμε στη συμβαστική Β που αφορά την παραγραφό 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Sì, όλε οι άλλε τροπολογίε και ψηφίζουμε τώρα το συμβασμό C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένω, καταπίπτουν οι άλλες. Τροπολογίες 25 και 26. 26 ψηφίσαμε. Να ψηφίσουμε την 26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωση. Δύο. Ποιοι είναι υπέρ. μετά αποχές απορρίπτεται. Καταθετεί το 3, το 4, το 5 και το 6. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και επομένω καταπίπτει το 7 και οι άλλε. <coughs> και πάμε τώρα στην συμβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα ε, κατευθείαν στο F, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε επομένω στην τροπολογία 43 του Λουί Μισελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται παράδειγμα το 44, πάμε στο 45, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 46, 47, ταυτόσιμες. Ψηφίσουμε ομού, υπέρ, κατά, αποχές. Α, απορρίπτεται. Βρισκόμαστε στο 3, παράγραφος 48. Όχι, τροπολογία 48 για τον κοντρά. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 52 μέχρι και το 54 που είναι ταυτόσιμες υπέρ Contrari. Κατά. Astenuti? Αποχές. Un astenuto, sono 10 favorevoli, 9 contrari. 19 E poi meno Επομένως εγκρίνεται.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 Votiamo. Emendamento 50. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Για να δούμε τώρα, ε, ε, έχουμε άλλε και πάμε στην ε, τελική ψηφοφορία. Όλο το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί, σηκώστε το χέρι. Υπέρ. 21 υπέρ, κατά, κατά, αποχές, 21 0 0. Ωραία, πολύ πολύ γρήγορα προχωρήσαμε, κάνουμε αυτή την πρώτη ψηφοφορία και πάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία. Αφορά το εξή. Το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία. Είστε έτοιμοι για να ψηφίσουμε. Πρώτη. Παράγραφος. Τροπολογία 14. Α, κύριε Ντάφη, για το λόγο. Νομίζω θα μπορούσαμε, αν συμφωνεί και ο κύριος Φόξ, να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες του ομάδας ECR μαζί. Όλες οι τροπολογίες ECR να ψηφιστούν μαζί. Αυτή είναι η πρόταση. Είμαστε υπέρ των περισσότερων, αλλά όχι όλων. Ποιε είναι οι τροπολογίε. Ε, καλά, καλά, τέλο Έτσι κι αλλιώ δεν είναι τόσο μεγάλη η ψηφορία. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Οπότε, ε, ας ψηφίσουμε μία-μία τι τροπολογίες. 14 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. Αριθμόν ένα, ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. προπολογία, τέσσερα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. πέντε, υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 8 υπέρ. Contrari. Κατά. Ε, Αστελού. Αποχές. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά 11-10. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Ο Ογιές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κοντράρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το ΕΡΤ, το, το που λέει 12 υπέρ. Κατά. Respinto. Astenuti. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τελική παραγραφός Η Καινούργια. Το 13. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Όταν μπορούμε να κάνουμε τελική ψηφορία. Υπέρ. Σηκώστε το χέρι. Αποχε... Κατά, κατά, κατά. Αποχές. Α, ε, εγκρίνεται. Εγκρίνεται και σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, επιτέλεσαν εξαιρετική δουλειά. Οι Ταρκόφσκη και Γουαλτιέρη συνεισηγητέ. Οπότε και τώρα. Allora c'è da dare le comunicazioni. Prima ακούσουμε τώρα τις ανακοινώσεις πριν κηρύξουμε την λήξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίστηκε όσον αφορά την Ερευνητική Επιτροπή αποφασίσαμε να συμμορφωθούμε με την ε, γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής και επομένως να μην τοποθετηθούμε κατά τρόπο διαφορετικό. Όσον αφορά δε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και την αναθεώρηση, έχουμε την πρόταση του Προέδρου και του εισηγητή. Όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό του 2014, θα οριστεί εισηγητής. Θα είναι ο κύριος Μέσες, εάν δεν υπάρχει ένσταση. Και όσον αφορά αυτό που ζήτησε ο συνάδελφος Νταφ, ε, θα κάνουμε την πρόσκληση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και όσον αφορά επίσης τα δικαιώματα των, ε, των βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης και όσον αφορά τώρα την αλλαγή, την τροποποίηση του άρθρου 100, συμμετοχή των βουλευτών στις ε, συνεδριάσεις. Είπαμε ότι η εισηγητής θα γίνει ο κύριος Χέφνερ. Oh, όσον αφορά το αίτημα του να συνταχθεί μια γνωμοδότηση Έτσι από την Επιτροπή Αναδείξης, είπαμε ότι δεν θα αλλάξουν, δεν θα αναθεωρηθεί ο κανονισμός. relazione sulla governance differenziata e, e poi infine. Eh, Τόσο αυτό ε, καλύπτεται όπως και άλλα θέματα από την έκθεση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα θα γίνει η ψηφοφορία. Όταν έρθει η ώρα επομένως να ψηφιστεί η έκθεση της κυρίας Γιαννέκου. Και είπαμε ότι θα γίνει αναβολή. 28 και 30 Μαΐου στο Λονδίνο θα συμμετάσχουν στην αποστολή αυτή 7 βουλευτές και βέβαια όσοι Βρετανοί θέλουν να συμμετάσχουν. Δύο από το ΕΛΚ, δύο από τους ε, ε, σοσιαλιστές και τρεις από τις ε, άλλες πολιτικές ομάδες. 7 και 8 Οκτωβρίου έχουμε συνεδρίαση με την Επιτροπή των Υποθέσεων και, και στη συνέχεια της απόφασης του δικαστηρίου. Οπότε και θα έχουμε μία συνεδρίαση στο Στρασβούργο, στην Ολομέλη. Οπότε και θα πάει για τότε η συνεδρίασή μας για 14 Οκτωβρίου τη Δευτέρα το απόγευμα. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Έχετε κάποιοι κάτι να παρατηρήσετε. Αποφασίσαμε επίσης ε, να παραμείνει η, ο, ο, ο τίτλος «Συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση απόσχησης». Λοιπόν, να παραμείνει η λέξη «απόσχηση». Σε περίπτωση απόσχησης, επομένως, κάποιου κράτους μέλους. Θα τα δούμε αυτά την επόμενη φορά και τη δικασία της επιλογής. Ευχαριστώ. Πέρασε συνεδριάσεις.